Γίνονται τα πρακτικά. Το πρώτο σημείο στην διάταξη είναι μια έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχές παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. Για τέσσερα λεπτά θα δώσω το λόγο στην συγκήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά συγκινημένη για το ότι σήμερα στην Ολομέλη αυτή θα ολοκληρώσουμε, ελπίζω, ένα φάκελο μακράς διαρκείας που έχει μια μακρά ιστορία και περιπετειώδη. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε καλό τέλος. Το 2008 υπό την Γαλλική Προεδρία μπορέσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή τη νέα πρόταση που συμπεριλάβανε αυτή την απόφαση να τεθεί τέλος ε, στην ατιμορρησία και να μειώσουμε την εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των παραβατών στον τομέα της ε, διασυνοριακή οδική ασφάλεια. Πρόκειται λοιπόν ε, για ένα διασυνοριακό ζήτημα που έχει και ω στόχο να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, να μειώσει τους τραυματίε και τα θύματα. Είναι αλήθεια όμως ότι το 2008 ξεκινήσαμε μία ε, τολμηρή και ολοκληρωμένη διαδικασία που βασιζόταν στις πληροφορίες ε, που είχαμε από τις οικογένειες των θυμάτων ε, σε οργανισμούς ευρωπαϊκούς ή και σε ενώσεις όπως η της ΠΟΛ που αφορούν την οδική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε οι διασυνοριακοί παραβάτες καταρχήν να ενημερώνονται για την παράβασή τους όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους και να μπορούσαν ε, να τους επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα έτσι ώστε να τεθεί τέλος στην ατιμορρησία. Όμως όπως τόσες φορές ε, δεν μας συνόδευσε το, δεν μας στήριξε το Συμβούλιο για διάφορους λόγους, μπλόκαρε την πρόθεση και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και να πατήσω φορτιμή στην ε, Βελγική Προεδρία που ε, μπόρεσε να αναστήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το φάκελο με μια άλλη νομική βάση της αστυνομικής συνεργασίας. Όμως ε, μπόρεσε και πάλι να θέσει σε τροχιά μια διαδικασία τόσο σημαντική για να θέσουμε τέλος στην ατιμορρυσία σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια και αυτή η Βελγική Προεδρία μαζί με την Ουγγρική ε, εκ νέου ε, εργάστηκαν υπό νομική βάση, αλλά μπορέσαμε να βελτιώσουμε κάποια σημεία. Χάσαμε την παρουσία σημαντικών κρατών μελών, όπως της Δανίας, Ιρλανδίας και του Βασιλείου, όμως μπορέσαμε αντί αυτού να βελτιώσουμε τον κατάλογο και βελτιώσαμε κάποιες από τις προτάσεις στα πλαίσια αυτής της αστυνομικής συνεργασίας, έτσι ώστε τον Νοέμβριο του 2013 Ήδη είχαμε ένα μέσο, ένα νομοθέτημα που ήδη δεν μπορούσε να μεταφορθεί στο ιστορικό δικαίωμα των κρατών μελών και εκείνη τη στιγμή, το Μάιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας ειδοποίησε για κάτι που είχαμε προβλέψει, ότι η αρχική νομική βάση που είχαμε προβλέψει η Κομισιόν και είχε υποστηρίξει το Κοινοβούλιο ήταν η βάση της οδικής ασφάλειας. Όμως αυτό προφανώς αποτελούσε ένα εμπόδιο τα κράτη-μέλη ήδη εφάρμοζαν και με καλά αποτελέσματα την οδηγία, ε, την ανταλλαγή πληροφοριών. Όμως ε, έπρεπε φυσικά να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο ήταν αρκετά ευφυές και μας άφησε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιους μήνες στη διάθεσή μας για να θέσουμε εκ νέου σε εφαρμογή το κείμενο και αυτό έκανε και η Κομισιόν και εκ νέου το Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρο και το τονίζω αυτό γιατί θα ήθελα να ζητήσω κάτι και από την Επίτροπο ΜΕΙΣ στο Κοινοβουλίο ε, θέλαμε ε, να ξανανοίξουμε την οδηγία γιατί η αρχική δεν μας άρεσε 100% Γι' αυτό θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, σήμερα να απευθώ σε εσά και να σας ζητήσω να προχωρήσετε όσο δυνατό ταχύτερα στην έκθεση αξιολόγησης και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι αυτό το φίλουμε στις οικογένειες των θυμάτων, ε, των δυστυχημάτων, ε, το φίλουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί μέσω τέτοιων νομοθετημάτων πρέπει να είναι ικανοί να πιστέψουν ότι πράγματι τους προστατεύει η Ευρώπη και μάλιστα σε κάτι τόσο σημαντικό όπως ε, είναι η απώλεια ζωή στο δρόμο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συγητρία η Επίτροπος Μπούλτς. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και ιδίως την κυρία Αγιάλα Σεντέρ, την εισηγήτρια, για την ταχύτατη εξέταση της εν λόγω πρότασης και την ολοκλήρωση της ε, έκθεσης εντός της προθεσμίας που έθεσε το δικαστήριο. Πρόκειται για τέλειο παράδειγμα πως ε, η καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων μπορεί να αποκομίσει ταχαία αποτελέσματα. Η Κομισιόν σας ευχαριστεί διότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα επί το οποίο επεφάθη το δικαστήριο πέρσι χωρίς να επεμπολίσουμε την αρχή της ε, αρχικής δηλαδή οδηγίας. Η νέα οδηγία θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια με βάση μάλλον την νομική βάση σε όλα τα κρατη τα 28 κρατη και όχι μόνο τα 25 όπως προηγουμένω, με νομική ε, βάση ε, που αφορά το των μεταφορών γιατί προηγουμένω είναι εξαιρετική η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Έτσι υπάρχει συνέχεια και θα βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια που είναι και ο βασικός στόχος, ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής μας στις μεταφορές. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός Ευρωπαίων γίνεται θύμα οδηγών που πολλές φορές δεν μπορούμε να εντοπίσουμε όταν να διαπράττουν παραβάσει σε άλλη χώρα μέλος. Πιστεύω λοιπόν ότι η οδηγία θα επηρεάσει από εδώ και πέρα την συμπεριφορά των οδηγών προς το καλύτερο. Διότι οι πολίτες μας αντιλαμβάνονται περισσότερο από ποτέ ότι η οδική ασφάλεια δεν σταματά στα εθνικά μας σύνορα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους μας πέραν των σύνορων. Η οδηγία αναφέρεται σε συγκεκριμένες παραβάσεις που όταν διαπράττονται θα είναι δυνατόν από εδώ και πέρα να εντοπίζεται ο οδηγός και το όχημα και θα ζητούμε από τον οδηγό εξηγήσει. Τέλος λοιπόν, στην ατιμορρησία των οδηγών σε χώρα άλλη από τη δική τους. Προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το απόγευμα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και ξεκινούμε με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Μπαχ καταρχάς για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχήν θέλω να ε, επενέσω για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Η οδική ασφάλεια αναμφίβολα είναι υψίστη προτεραιότητά μας. Μόνο με κοινέ και διασυνοριακές προσπάθειες θα μπορέσουμε ως το 2020 να μειώσουμε κατά το ίμιση των νεκρών στην άσφαλτο και ε, βεβαίως εδώ χρειάζονται μέτρα εκπαίδευσης, καλύτερη υποδομή, σύστημα ασφάλειας μέσα και έξω από τα οχήματα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη οδική ασφάλεια. Πολύ σημαντικό είναι ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμόζεται και στα 28 κρατή-μέλη και στις 3 ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία και ήδη 20 χώρες την έχουν ε, ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο. Οι υπόλοιποι ελπίζω ότι θα κάνουν κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να τηρήσουν την προθεσμία ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Σημαντικό είναι οι οδηγοί να ε, αντιμετωπίζονται ισότιμα, είτε η μεδαπή είτε αλλοδαπή. Όλοι θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις. Ε, αν ε, είναι, οδηγούν πιωμένοι, υπερβαίνουν τα όρια ε, ταχύτητας, το όριο ταχύτητας, θα πρέπει να τιμωρούνται το ίδιο. Χρειάζεται γι' αυτό αναπροσαρμογή των δεδομένων και της προστασίας των δεδομένων. Εδώ προσέξαμε ιδιαίτερα το θέμα. Η οδική ασφάλεια, η ασφάλεια των μεταφορών ε, χρειάζεται προσπάθειες από όλους γιατί ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς σε ορισμένες χώρες ε, αυξάνονται πάλι. Εγώ είμαι αισιόδοξο και όπως είπε και η συνάδελφος Αγιάλα Σέντερ, ε, είμαι αισιόδοξο ότι η Κομισιόν μέχρι το Νοέμβριο του 2016 θα αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις και θα υποβάλει την έκθεση. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ε, αντιμετωπίσουμε τα καθήκοντά μας και θα ανταποκριθούμε σωστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ερτούκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, τουλάχιστον μπορέσαμε να απαντήσουμε στο αν αυτοί που κάνουν αδικήματα στο εξωτερικό, αν αυτοί μπορούν να διωχθούν ε, στο συνολικό μόρφωμα των 28. Δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα. Μην ξεχνάμε όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ε, αν ε, δούμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής μηδενικής ανοχής ε, βλέπουμε ότι έδωσε καλά αποτελέσματα και μειώθηκε ο αριθμός των θυμάτων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τώρα όταν ε, δημιουργηθεί θέμα σε ένα κράτος μέλος, τώρα μπορεί να ε, ενημερωθούμε. Μετά όμως τι θα γίνει. Ε, αυτό απασχολεί τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Η εκτέλεση, δηλαδή η ίσπραξη του προστίμου δεν επιτυγχάνεται. Αν υποθέτουμε δηλαδή ότι αυτός ο οποίος έκανε την παράβαση άρνητα να πληρώσει το πρόστιμο. Σε αυτή την περίπτωση και το λέω συνειδητά αυτό γιατί ξέρω ότι το 2016 πρέπει να κάνετε μια αξιολόγηση. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει στην επόμενη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν να τα ε, αναφέρετε και να τα ρυθμίσετε γιατί μόνο τότε θα έχουμε ρυθμίσει σωστά το θέμα μας. Αν ξέρει ο παραβάτης ότι δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο. Είναι πολύ καλή η προσπάθεια. Ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια για την καλή δουλειά και προσβλέπω στη νέα νομοθετική πρόταση που θα τα ρυθμίζει όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Βαντάλεν, δύο λεπτά. Πρόεδρε, κάθε χρόνο 25.000 πολίτες μπλέκονται σε ατυχήματα και αν ε, λάβουμε υπόψη και τους ε, πολίτες ε, που δεν βρίσκουν το θάνατο αλλά παραμένουν αναπερίτωτοι, θα έχουμε ένα νούμερο συγκρίσιμο με τον πληθυσμό μιας ολόκληρης χώρας. Μπορούμε να έχουμε φύγει οχήματα, καλύτερη υποδομή και καλύτερες πληροφορίες και καλύτερη παροχή βοήθειας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα. Η Κομισιόν ξεκίνησε ε, νομικές διαδικασίες κατά του Συμβουλίου, όμως εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε ένα επίγον κοινωνικό ζήτημα. Όμως ε, ελπίζω ότι με την έγκριση αυτής της πρότασης θα βρούμε μια λύση και θα προωθήσουμε την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Είναι τώρα πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε τις τροχές παραβάσεις για συνοριακού χαρακτήρα, ιδίως όταν μιλάμε για ε, κάποιες παραβάσεις ε, όπως το να οδηγεί κανείς υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ ή την υπερβολική ταχύτητα. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι η κατάσταση. Ελπίζω ότι δεν θα μείνει όλη αυτή η πρωτοβουλία στα χαρτιά. Λέγεται ότι θα δοθεί και ενημέρωση ε, στους οδηγούς. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει όλοι να ενημερώνονται σωστά, έτσι όλοι να γνωρίζουν ότι πρέπει να οδηγούν υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μπιλμπαμπεραντίκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Ο Παγκοσμίο Οργανισμό Υγεία υπενθυμίζει στι μελέτε ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι ο έβδημο λόγο ε, θνησιμότητα ε, στον ε, κόσμο και θα, το 2030 θα είναι ο πέμπτο λόγο αν δεν μπορέσουμε να μειώσουμε τα ατυχήματα αυτά. Πρέπει να προωθήσουμε την ε, χρήση ε, της ζώνης ή του κράνους, να μειώσουμε την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, ε, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δυστυχημάτων η οδηγία που συζητούμε σήμερα θέλει να βελτιώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Η αλλαγή τη νομική βάση θα επιτρέψει Δανία, Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή στην εσωτερική του νομοθεσία. Το να επιτρέψουμε ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ των κρατών σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση των οχημάτων τη Ευρώπη ε, και να μπορούμε να τιμωρούμε όλους τους παραβάτες ανεξάρτητα με το που έχει γίνει η παράβαση των κανόνων οδικής ασφάλειας. Επίσης, ελπίζω ότι θα προωθηθεί συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και έχουμε αποκεντρωμένες αρμοδιότητες στο τομέα αυτό επίσης. Θα, μειωθεί, θα μειωθούν τα δυστυχήματα σε όλη την Ευρώπη γιατί έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα παρά όλα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς κατανέμονται τα θύματα και τα δυστυχήματα εντός των κρατών μελών. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης οι χώρες με τα περισσότερα ατυχήματα θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τις υποδομές, για το στόλο των αυτοκινήτων και άλλα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγουμε να έχουμε 55 νεκρούς ε, για ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Το 2017 η Κομισιόν θα μας ε, παρουσιάσει μία νέα πρόταση με νομική βάση ε, στις μεταφορές και ελπίζουμε να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κιλιόνεν. Συνάδελφοι, μία κοινή, ένας κοινός χώρος μεταφορών απαιτεί μια τέτοια οδηγία, σαν αυτή που συζητούμε σήμερα. Κοινοί κανόνες λοιπόν σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο εναντί όλων. Είναι ένας μηχανισμός αποτροπής για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητος του αν διαπράττουν μια παραβάση στη μία την άλλη χώρα. Είναι θέμα δικαιοσύνης, ισότιμης μεταχείρισης, από τις πλευράς του νόμου και αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και το Συμβούλιο διότι επιτάχυναν τις σχετικές συνομιλίες. Ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε και εμείς εδώ το κείμενο ώστε να υπάρχει απόλυτη νομική σαφήνεια και βεβαίως να γίνουν και τα επόμενα βήματα ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς η υπερβολική ταχύτητα, η άγνοια της ε, υποχρέωσης εφαρμογής της ζώνης ασφαλείας, ε, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Είναι βασικές αιτίες θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατοντάδες θα μπορούσαν να σωθούν με τη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Ευχαριστώ. Κύριος ένα λεπτό από τους πράσινους. Κυρία Πρόεδρε, πρώτον να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πραγματικά για το έργο σας. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα την προσπάθεια όλων ε, δεν ξέρω αν ήταν υποδηματική η συνεργασία μας, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο. Χάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας την νομική βάση και είναι κρίμα που το Συμβούλιο αναλώθηκε σε μια τέτοια γενική συζήτηση, αλλά επιτέλους τώρα πια μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Οι σχετικές διατάξεις είναι ικανοποιητικέ. Ας ασχοληθούμε πλέον με την εφαρμογή, με την ε, ενσωμάτωση και μετά εφαρμογή της οδηγίας της Εθνικής Ένωμες Τάξης. Γιατί μέχρι την αναθεώρηση του 2016 πρέπει να έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε την οδηγία για να βελτιώσουμε τις συνθήκες, τους δρόμους της Ευρώπης. Δεν ήταν ιδανική λοιπόν η συνεργασία, αλλά τέλος πάντων τελειώσαμε με αυτά και μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας πια το 2016. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντγκρεν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες, γιατί δεν λειτουργούν καθοδόν καλά. Πολλές φορές αλλοδαποί είναι πεπισμένοι ότι μπορεί να γλιτώσουν οποιοδήποτε πρόστιμο τους επιβάλλει η αστυνομία. Δεν υπάρχει σύστημα που θα εισπράξει τα πρόστιμα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στην έκθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχουν έλεγχοι των οδηγών, έλεγχοι της κυκλοφορίας με ένα σύστημα αναλογικό. Αυτό είναι πολύ σωστό και πρέπει να υποστηρίξουμε την αστυνομία που κάνει σκληρή δουλειά για να τους ελέγχει. Ή τα πρόστιμα ή δυνατόν πρέπει να καταβάλλονται επί τόπου, γιατί αλλιώς όλο και θα ξεκλειστρούν από το δίχτυ. Δηλαδή μια εταιρεία μεταφορών, ας πούμε, γιατί να μην έχει μια πιστοτική κάρτα στους οδηγούς της για να πληρώνουν τα πρόστιμα. Με αυτήν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ρυθμίσουμε. Επίσης ε, τα πλαστά διπλώματα οδήγησης θα πρέπει να τα πιάνουμε γιατί πολλές φορές τα αγοράζουν ε, από το διαδίκτυο και, ε, δεν, και, έχουν επαγγελματικά που δεν δικαιούνται. Αυτό πρέπει επίσης να το ρυθμίσουμε. Κυρία η οδηγία αυτή επιστρέφει στην Ολομέλεια ε, ότι όταν ε, πρόκειται για δίωξη ε, των οδηγών κάποιοι που μένουν εδώ φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσουμε τις παραβέας του ΚΟΚ είναι η δίωξη των οδηγών σε ό,τι αφορά την ε, ανανέωση του δικού δικτύου και την ε, συντήρησή του θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ποτέ φυσικά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε γιατί ε, κοστίζει πολλά ενώ τα ραντάρ είναι πολύ ωφέλιμα σε ό,τι αφορά κάποιους αμυντές που συχνά οδηγούν κλεμμένα οχήματα τίποτα δεν λένε ξέρετε το περασμένο μήνα είχαμε κάποιους ε, που προκάλεσαν ένα θανατηφόρο δυστύχημα ε, και δεν είχαν ούτε άδεια ούτε ταυτότητα. Πιστεύετε ότι αυτή η οδηγία θα μας επιτρέπει να ε, καταπολεμήσουμε το αδίκημα του GoFast Από ό,τι φαίνεται όχι. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει κάποια ευελιξία για τους κανονικούς οδηγού, αλλά να υπάρχει και μηδενική ανοχή για τους εγκληματίες του δρόμου. Mr. Van de Κύριε Σουαντεκάμπ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο θέμα ο κύριος ε, Βαντάλεν είπε ότι 25.000 ε, φωνεύονται στον δρόμο κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Φρικτό νούμερο. Πρέπει να κάνουμε το παν για να μειώσουμε τον αριθμό αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Εμείς στην ομάδα μας πιστεύουμε ότι είναι καλό να κλείσουμε το φάκελο αυτό σήμερα με μια ξεκάθαρη ψήφο υπέρ. Προφανώς όταν μιλάμε για διασυνοριακές ε, τροχές παραβάσεις ε, θα έχουμε, ε, τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όμως δεν θα είναι τόσο εύκολο να θεωρεί ο κάθε ένας ότι μπορεί να γλιτώνει από τα πρόστιμα. Ε, μπορεί κάποιοι να γλιτώνουν, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για τροχές παραβάσεις, φαντάζομαι επικεντρωνόμαστε στις πιο σημαντικές και σοβαρές. Ε, η Γερμανία, κάτω χώρες, ε, Βέλγιο ανταλλάσσουν για παράδειγμα περισσότερες πληροφορίες και για άλλες τροχές παραβάσεις. Α, Τώρα, για την ε, εφαρμογή ε, και την επιβολή των μέτρων ε, έχουμε έτοιμα τα μηχανογραφικά συστήματα σε όλα τα κράτη-μέλη και μπορούν να είναι διαλειτουργικά. Γιατί πολλές φορές είχαμε σφάλματα που οφείλονταν στους υπολογιστές. Καλό είναι ότι οι τρεις χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, θα συμμετέχουν σε ισότιμη βάση. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά η κυρία Άντερσον. Εγώ το χαιρετίζω ιδιαίτερα το μέτρο αυτό και την υποστήριξη της, ε, που δίνουμε στην Επίτροπο. Μην κάνουμε λάθος. Αυτό είναι μέτρο δικής ασφάλειας. Είναι για την αποτροπή και την καλή διακυβέρνηση. Δεν είναι για επαχθείς ε, και άδικες ρυθμίσεις όλα αυτά είναι σοβαρά, σοβαρές ε, παραβάσεις. Ιδιαίτερα η υπέρβαση του ορίου ταχύτητος είναι ε, υπεύθυνη για περισσότερο από το 1 τρίτο των θανατηφόρων τροχαίων και επιβαρύνει την κατάσταση σε άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να το θέσω υπό έλεγχο. Στη χώρα μου ξέρω ότι δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτό η πρόταση. Πολλές φορές ε, προσπαθήσαμε να ε, κρατηθούμε απ' έξω. Εγώ καλώ την κυβέρνησή μου να αλλάξει άποψη και να προσπαθήσει να τα εφαρμόσει ταχύτερα όλα αυτά από ό,τι υποσχέθηκε. Τώρα για τα στοιχεία τα αριθμητικά υπάρχουν πολλά ακραία στοιχεία για το πώς μπορούμε να ε, τα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, στο περιφερειακό του Λονδίνου έχουμε ε, στοιχεία πολύ ανησυχητικά και στην που ε, και οι παραβάσεις στον ε, περιφερειακό στο Λονδίνο ε, πολλές παραβάσεις γίνονται από ξένους οδηγούς. Το ίδιο ισχύει και στην Γαλλία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερα πράγματα για να επιτύχουμε τους στόχους οδικής ασφάλειας το 2020 όπως έχουμε θέσει. Και θα πρέπει οι όροι για την οδική ασφάλεια να ε, ληφθούν υπόψη και στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεταφορές ε, και για την, ε, τις μεταφορές. Η οδική ασφάλεια θα πρέπει να θεωρείται πάντοτε μια κορυφαία προτεραιότητα. Έχετε, υπάρχει μπλε κάρτα. Ποια, ποιον, για την κυρία Άντερσον η ερώτηση. Ναι, Δέχεστε από τον κύριο Ρόπερ τη μπλε κάρτα. Ναι, κύριε Ρόπερ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανταλλαγή των ε, πληροφοριών θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τον αριθμό των παραβάσεων, αλλά με ενδιαφέρει το εξής, αν η δεσμευτική απέτηση να οδηγεί ε, κάποιος ε, ε, όταν το τιμόνι είναι δεξιά είτε αριστερά, αυτό μήπως θα υποσκάψει την νομοθεσία. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον τύπο του οχήματος, χωρίς μικρόφωνο. Κοιτάξτε, το εξετάζουμε αυτό το θέμα πολύ λεπτομερώς στη χώρα μου. Ε, αλλά και σε άλλες για να διασφαλίσουμε ότι από τεχνική σκοπιά όταν ε, ε, έχουμε να κάνουμε με θέματα υποδομής και με μέτρα. Λαμβάνουμε υπόψη και την οδική ασφάλεια για τα οχήματα που έχουν το τιμόνι από την άλλη πλευρά. Και Επίσης ε, αυτό το έχει κατά νου και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η υπηρετική Ευρώπη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με θέματα οδικής ασφάλειας το έχουμε κατά νου. Μάλιστα, επόμενος ε, ομιλητής, ο κύριος Σλοτόφσκι, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ η ε, ελευθερία Μετακίνηση και η κυκλοφορία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα κύρια κεκτημένα. Αλλά το προνόμιο όσων κινούνται στους οδούς της Ευρώπης ε, σημαίνει ότι ε, θα πρέπει ε, να είναι απολύτω υπεύθυνοι για τις παραβάσεις, να λογοδοτούν για τις παραβάσεις και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα κατάλληλα μέσα για να καταπολεμά τις παραβάσεις του κωδικού κυκλοφορίας. το να επικαλείται κάποιος ότι δεν γνωρίζει την διεύθυνση του παραβάτη είναι μια δικαιολογία που δεν μπορούμε να τη δεκτούμε στην Πολωνία. Ο ρυθμός των δυστυχημάτων είναι πάρα πολύ υψηλός και η ενορμόνιση αυτών των διατάξεων μας ικανοποιεί ιδιαίτερα στην Πολωνία. Περίπου 3% όλων των συγκρούσεων και των ατυχημάτων στο δρόμο είναι ατυχήματα που δημιουργούνται από αλλοδαπούς και κυρίως από Ευρωπαίους πολίτες. Φυσικά κάθε δυστύχημα είναι τραγικό και η δυνατότητα να τιμωρηθεί ο παραβάτης ε, σίγουρα έχει και εκπαιδευτική αξία. Θα πρέπει να ε, τονίσουμε ότι οι τριτές χώρες που μέχρι ε, τώρα αποκλείονταν από το σύστημα είναι τώρα έτοιμες να μπουν. Πρέπει το σύστημα αυτό να καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη και είμαι πολύ ικανοποιημένο που πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν θέσει αυτές τις διατάξεις σε εφαρμογή. Θα ήθελα επίσης να φυστήσω την προσοχή σας στο εξή ότι θα ήταν χρήσιμο να διευρύνουμε τη διάταξη αυτή για να καλύπτει και τις όμορες χώρες. Ο κύριος Ρικέ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, τη συναδελφή, συγχαρητήρια στην κυρία για το έργο της που οδηγεί σε μια νέα οδηγία στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο. Θα βελτιώσουμε την ασφάλεια στους δρόμους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία 21% των παραβάσεων ε, το κόκκινο και η περιβολική ταχύτητα οφείλεται σε οδηγούς από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν αποκαθιστούμε ισότιμη μεταχείριση μεταξύ όλων των παραβατών για τα δικήματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Είναι ενδεχομένω το πρώτο βήμα για να επικρατήσει επιτέλου ένα κώδικα καλή οδική συμπεριφορά στην Ευρώπη. Φυσικά εκκρεμούν ορισμένα ερωτήματα. Τι θα γίνεται, για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιο δεν πληρώνει το πρόστιμο, πώ ε, εφαρμόζονται οι κυρώσει, πώ συνεργάζονται τα κράτη-μέλη κλπ. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε το 2016 για να γίνουν οι απαραίτητε προσαρμογέ για την εκτέλεση και εφαρμογή των κυρώσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Σέιμου, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το νομοθέτημα δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη εξαιτία τις επικαλυπτόμενες νομοθεσίες. Δυστυχώ, ακόμη και σήμερα μετά την οδηγία πριν δεν έχουμε τα στοιχεία, του τύπου δεδομένων που χρειαζόμαστε για την οδική ασφάλεια. Δύσκολα θα εφαρμοστεί λοιπόν μια τέτοια οδηγία, φοβούμε, γιατί η αστυνομία δεν έχει τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να τιμωρήσει του παραβάτε. Πρέπει λοιπόν στα σύνορα να καταχωρούνται τα στοιχεία, οι πινακίδες των αυτοκινήτων και οι άδειε των οδηγών. Έτσι, όταν θα βγαίνει κανείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, θα μπορεί η αστυνομία να τον σταματάει και να τον τιμωρεί αρμοδίως. Χρειάζεται λοιπόν να τυποποιηθούν οι τεχνολογίες στα σύνορα, τεχνολογίες ελέγχου. Το γλωσσικό θέμα δεν είναι πρόβλημα. Φοβούμαι όμω εν τέλει ότι η οδηγία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Ο αρμόδιο Άγγλος Μεταφορών είπε επίση ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα σημείων, ένα point system. Αυτό καλό θα είναι να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. οι βουλευτέ του UKIP θέλουν να προστατεύσουν πραγματικά τα συμφέροντα των οδηγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει μια μπλε ε, κάρτα όμω από ό,τι βλέπω. Κύριε Σέιμορ, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρτη. Ε, παρακαλώ κύριε Κάρτη. Τα επιχειρήματά σα θα είχαν νόημα εάν η χώρα σας δεν έχει αρμοδιότητα για τμήμα της χώρας που εκπροσωπώ. 500 δρόμοι στην Βόρειο Ιρλανδία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Δεν ε, συμφωνείτε ότι πρέπει με ένα κάποιο σύστημα να μπορούμε να καθιστούμε τους οδηγούς υπεύθυνους και από την άλλη πλευρά των συνόρων. και Ναι, φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, αλλά είναι αρμοδιότητα δική μας εθνική και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία. για να μισή Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια στους δρόμους μας είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Αυτό προκύπτει από αυτά που ακούσαμε διαπαραταξιακά. Ισχύει αυτό. Η Αυστρία πλήττεται από τα προβλήματα αυτά. Ε, ιδιαίτερα από τη μεταφορά Ανατολή προς Δύση. Οπότε τα μέτρα είναι ευπρόσδεκτα. Ε, τα από 4 εκατομμύρια παραβάσεις, τα 2,5 ε, όπως εντοπίζονται από τον ραντάρ, γίνονται από ξένους. Σημαντικό είναι η εφαρμογή βέβαια της οδηγίας όπως ξέρετε όλοι. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν εφαρμόσει η Ιταλία, η Ελλάδα αναφέρθηκαν ότι δεν είχαν εφαρμόσει την προηγούμενη οδηγία και από την άλλη το θέμα είναι αν όλα τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα και αποτελεσματικά μπορούν να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. Το πρόβλημα της διοίκησης επίσης αναφέρθηκε για κάποια κράτη. Πάντως, παρόλα αυτά, οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους, δηλαδή τα κράτη-μέλη όλα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή, διότι οι πολίτες των χωρών που θα εφαρμόσουν καλά την οδηγία θα είναι ε, ε, εκείνοι οι πολίτες που θα πληρώνουν πιο πολύ τα πρόστιμα. Ε, αν δεν τα κάνουμε σωστά. Ο κύριος Κοχ, δύο λεπτά. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι πολύ μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που μας ενδιαφέρει στην τεράστια πλειοψηφία μας. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται βαριά μετά από παραβάσεις. Οι παραβάσεις, ε, οι σοβαρές μας είναι πολύ γνωστές, είναι υπερβάσεις ορίων ταχύτητας, η μέθη στο τιμόνι, η ε, οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ε, μη χρήση, η παραβίαση του κόκκινου, ε, μη χρήση ζώνης. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται το όχημα, σε ποια χώρα θα πρέπει να τιμωρείται. Οι σοβαρές τροχές παραβάσεις δεν μπορεί να μην διώκονται σε μια οργανωμένη ε, χώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι μπορούμε και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δεδομένων να έχουμε πρόσβαση ε, στη, στα στοιχεία του οδηγού. Αυτό διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία ε, επίδοσης του προστίμου στον παραβάτη. Ε, έχουμε και από το Μάιο του 2014 την απόφαση του δικαστηρίου που με καθησυχάζει. Δεν υπάρχει πια ε, εξαίρεση των χωρών Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία. Δεν μπορούν να αρνηθούν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Η οδική ασφάλεια δεν θα σταματά στα χερσαία σύνορα. Ε, η, άλλωστε η κινητικότητα των πολιτών έχει γίνει ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Τώρα θα πρέπει να ε, μην επαναπαυθούμε σε αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα, αλλά να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμόντε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση που εξετάζουμε ε, αναφέρεται στην οδηγία 12-2011 που ακυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί είχε λαθασμένη νομική βάση. Τώρα κάνουμε ένα νέο βήμα προς τον πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γιατί διευκολύνεται η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα οδικής ασφάλειας όπως φέρνουν χάρη την ε, υπερβολική ταχύτητα και θέτει τέλος ε, στην ατιμορρησία των μη διαμενόντων οδηγών. Ε, αυτό θα μας ε, οδηγήσει να αποδείξουμε ότι όλοι οι οδηγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Θα πρέπει οι κανόνες να γίνονται σεβαστοί από όλους. Ως, θα λαμβάνουν όλη ε, την παράβαση γιατί ανεξάρτητα που έχει ταξινομηθεί το όχημα ε, σε όλους ε, θα στέλνετε το πρόστιμο. Έτσι υπάρχει και η δυνατότητα να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τις άλλες χώρες και θα βελτιωθεί η ασφάλεια αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τέλειωσε λοιπόν η εποχή τη ατιμορρησία και νομίζω ότι ένα βήμα προ τα μπρο θα ήταν να επιτρέψουμε όχι μόνο την ανταλλαγή πληροφορίων αλλά και τη δυνατότητα να εφαρμοστεί απευθεία η κύρωση. Θα ήταν λοιπόν επιθυμητή μια αναθεώρηση τη οδηγία και προ αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σήμερα υπάρχει μια αλλαγή τη νομική νομικής βάσης και αυτό δεν είναι μόνο τυπικό αλλά είναι και ουσιαστικό στοιχείο για να ευαισθητοποιήσουμε του πολίτε ε, για την οδική ασφάλεια και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μάισνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μέχρι τώρα υπήρχε ατιμορρησία στην περίπτωση αυτή. Αλλά αυτό είναι ανεπίτρεπτο πλέον. Εμείς έχουμε φροντίσει με προσαρμογή στο σύστημα επιθεώρησης των ε, οχημάτων και τώρα βέβαια και διασυνοριακά ε, ε, διώκουμε τους παραβάτες. Είναι σημαντικό να παίρνουν στοιχεία τα άλλα κράτη-μέλη για τους παραβάτες. Η κινητικότητα είναι πολύ καλό πράγμα, αλλά θα πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες που θα τηρούνται από όλους. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι έχουμε το θέμα πάλι στην ημερήσια διάταξη, ούτω ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες νομικές προσαρμογές που θα επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση, χωρίς όμως ατιμορρησία των σοβαρών παραβατών. Θέλουμε ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης και στηρίζουμε την Επίτροπο ε, κατά την προσπάθεια εφαρμογής οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το ότι ξαναβλέπουμε αυτό το έργο δεν μας, μας απαγορεύει να αναφέρουμε ε, τον κύριο Μπουελά. Έχουμε ένα ολοκληρό πρόγραμμα όταν μιλάμε για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ε, κάτι θα μπορούσε να μεταφραστεί ως πίνουμε νερό κτλ. Τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ουσιαστικά μας ξαναστέλνει αυτή την οδηγία γιατί είχε υιοθετηθεί με λανθασμένη νομική βάση αλλά διατηρεί το ίδιο σκεπτικό. Εδώ θέλουμε να διώξουμε τα πιο, τις πιο σοβαρές ε, παραβάσεις ε, του ΚΟΚ. Φυσικά συμφωνώ, αλλά μεταξύ αυτών των παρεμβάσεων έχουμε παραδείγματος χάρη και το ότι κάποιος δεν έχει δέσει τη ζώνη ασφαλείας και φυσικά αυτό θέτει σε κίνδυνο ε, την ε, ε, ζωή του οδηγού αλλά όχι του άλλου. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δεν καλύπτονται με συγχωρείτε από αυτή την οδηγία ε, και ήδη ασχολούμαστε εδώ και τέσσερα χρόνια με αυτό το ζήτημα το Λουξεμβουργό, το οποίο έχει συνυπογράψει την συνθήκη του ΠΡΙΜ. Έπρεπε να μεταφέρουμε στο εσωτερικό δικαιώμα σε αυτή την οδηγία, όμως ε, ξέρουμε το χάρη ότι ε, κάποιοι απατεώνες στο δημόσιο τομέα μπορούσαν να δρούν ατιμόρυτα. αν θέλουμε εδώ τώρα να ελέγξουμε τις σοβαρές παραβάσεις, ναι, αν ε, θέλουμε τώρα εδώ να υιοθετήσουμε ένα μηχανισμό που απλώ ε, θα τιμωρεί τους οδηγούς, όχι, δεν συμφωνούμε. Η κυρία Κλούν. Βεβαίω να υπάρχει μια νομική βάση και να μην υπάρχουν κενά για να τιμωρούνται αυτοί που διαπράττουν παραβάσεις στη μία και την άλλη χώρα. Τέρμα λοιπόν στα τιμωρησία των οδηγών. Αυτό πρέπει να αλλάξει σήμερα και βεβαίω συμφωνώ. Η οδηγία πάνω απ' όλα αφορά την ασφάλεια. Και χαιρετίζω το γεγονό ότι πέρασε η έκθεση από την Επιτροπή μα την Επιτροπή Μεταφορών, στα οποία είμαι μέλο και ευχαριστώ και τη Σκιώδη Συγκήτρια και τον κύριο Μπαχ για την συνεργασία του. Έχουμε λοιπόν νέε προτάσει οι οποίε θα περιορίσουν τα θύματα των τριχιών ατυχημάτων κατά 300-400 το χρόνο. Αυτά δείχνουν οι μελέτες. Πέρα από τους ε, τρομερούς τραυματισμούς που επίσης ε, έχουμε στους δρόμους μας. Όμως, πέραν αυτών, θα βοηθήσει η οδηγία να σώσουμε περισσότερες ζωές, όπως είπα, στους δρόμους και να λειτουργήσουμε ως μια ενιαία Ευρώπη. Δεν γίνεται να ισχύουν δύο διαφορετικοί κανόνες για αυτούς που οδηγούν από τη χώρα μας και τους ξένους. μεταξύ των παραβάσεων. Το θέμα της ε, ζώνης είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει μάλιστα οι ενήλικοι να φροντίζουν τα παιδιά να φορούν ζώνη σε κάθε περίπτωση. Σημαίνει λοιπόν σημαντική πρόοδος και ξέρω κύριε Επίτροπε ότι είναι προτεραιότητά σας να μειώσετε τον αριθμό των θανάτων στου δρόμους μας. 76.000 άνθρωποι πέθαναν πριν από λίγα χρόνια στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ε, το κατεβάσαμε το νούμερο στο 26.000 αλλά Ακόμη το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. Προσβλέπουμε λοιπόν και στη δική σας συμβολή κύριε Επίτροπε τα επόμενα χρόνια για να μειώσουμε ακόμη τους θανάτους και να βελτιώσουμε τις συνδίκες ασφαλείας στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Κύριε Λουκασιεύσκα, 1,5 λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, ζητάει πρόεδρος. Η κυρία Σενάλοβα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ στην κυρία Γιάλα Σεντάρ, στη συνάδελφο, γιατί ολοκλήρωσε επιτυχώ το έργο τη γρήγορα. Ένα εξαιρετικό έργο σχετικά με μια οδηγία που είναι πολύ σημαντική, την οδική ασφάλεια. Αποτελεί όμως και το επιστέγασμα πολιτών προσπαθειών για να εφαρμοστεί μια τέτοια νομοθεσία επιτέλους στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου Έγινε άλλο ένα βήμα προς την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η οδηγία θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να περιορίσουμε το πλήθος των θανάτων κατά 50% στους ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 2020. Ευτυχώς τώρα πια έχουμε μια οδηγία η οποία επικεντρώνεται στις σημαντικές παραβάσεις, στην περιβολική ταχύτητα, την οδηγία από την εμπειρία αλκοόλ, ναρκωτικών και ούτω ε, την χρήση μεταξύ άλλων βεβαίω των κινητών τηλεφώνων, την παραβίαση του έρθρου σηματοδότη, ε, την οδήγηση με τους χωρίς δίτροχου, χωρίς κράνος κλπ. Χάρη στην οδηγία θα έχουμε πλέον ισότιμη μεταχείριση όλων των οδηγών σε όλους τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι οδηγοί θα γίνουν πιο υπεύθυνοι και θα προστατεύονται καλύτερα και αυτοί οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε ατυχήματα. Τέλος λοιπόν και στην ατιμωρήσια. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σα. Κυρία Λουκασίευσκα, Ευχαριστώ πολύ. Η ατιμορρησία των αλλοδαπών οδηγών είναι ένα πρόβλημα που συζητούμε εδώ και πολύ καιρό σε διεθνές επίπεδο. Οι κυβερνήσει, τα μέσα μαζική ενημέρωση και οι πολίτε συχνά το συζητούν. Κανένα δεν είναι ευχαριστημένο με τη σημερινή κατάσταση. Τα στατιστικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι οδικέ παραβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύουν ότι εκατοντάδες, ε, ακόμη και χιλιάδες ε, διαπράττουν τέτοιες ε, παραβάσεις και μάλιστα οι μη διαμένοντε, ε, τέτοιοι οδηγοί είναι περισσότεροι από του διαμένοντε. Έχουμε πάρα πολλού ανθρώπου που χάνουν τη ζωή του ε, στο δρόμο κάθε χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι ακόμη και η καλύτερη νομοθεσία δεν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική αν ο οδηγός ε, πιστεύει ότι είναι ατιμόρυτος. Ορισμένα άτομα μπορούν να παραβιάζουν καθημερινά διάφορους κανόνες ε, στην επικράτεια ενός άλλου κράτου όταν ξέρουν ότι δεν θα τους συμβεί τίποτα. Εγώ χαιρετίζω λοιπόν αυτή την οδηγία για την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύω ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα μειωθεί η ατιμορρησία και όλοι οι οδηγοί θα αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εθνικότητά τους. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω αυτή την οδηγία και ευχαριστώ την εισηγήτρια διότι αφενός Θέλουμε ε, όλο και περισσότερη απασχόληση, καλύτερη δημογραφική εξέλιξη. Ε, από την άλλη, 20.000 άνθρωποι ετησίως χάνουν τη ζωή τους ε, στις, ε, στους δρόμους της Ευρώπης. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να μένουν ατιμόρυτοι οι παραβάτες. Γι' αυτό είναι μια ρύθμιση οδηγία αυτή η οποία έρχεται ε, σε πολύ σωστή στιγμή. Υπάρχει και ε, φροντίδα για την απλοποίησή τη και είναι θετικό βέβαια ότι προσχωρούν και οι τρεις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία. Μέχρι το 2020 θα φροντίσουμε λοιπόν ώστε να μειωθούν κατά το ίμιση ε, τα θύματα στους δρόμους Όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Όμως η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ναι μεν είναι καλή, αλλά η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών δεν είναι πάντα τόσο εξαιρετική. Εκεί πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Αυτό ανταποκρίνεται και στην ευρωπαϊκή ιδέα. Σίγουρα οι κυρώσεις δεν είναι πανάκια, χρειάζεται καλύτερη υποδομή, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερα οχήματα και όλα αυτά τα μέτρα από κοινού θα ε, φροντίσουν να, βελτιωθούν, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Τα εθνικά σύνορα δεν είναι πια πραγματικά σύνορα και αυτό έχει πολλά θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε με το Catch the Eye. Η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για παραβάτες ε, τροχαίους ε, ξεπερνά την απλή αστυνομική συνεργασία ε, και αυτό αποτελεί θέμα ασφάλειας που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή εδώ η οδηγία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων που πρέπει να υποδιπλασιαστούν μέχρι το 2020. Αυτή είναι μια αποστολή που έχουμε αναλάβει, ένα καθήκον μας απέναντι στους πολίτες που μας έστειλαν εδώ. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι χρειάζεται βελτίωση, χρειάζονται βελτίωση υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε πάνω στην έννοια της ελεύθερης διακίνησης ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο προσώπων ε, αλλά και διασυνοριακή επικοινωνία εν προκειμένου για τους τροχαίους παραβάτες. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έχει σχέση με την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Απαιτείται λοιπόν να θεσπιστεί μια νέα νομική βάση για την οδηγία για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις. όπως προκύπτει από μελέτες των δεδομένων σε σχέση με τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και τις παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας το ποσοστό των μη κατοίκων που εμπλέκονται ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο των κατοίκων. αυτό μάλιστα αφορά ιδίως την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ο μεγάλος αριθμός παραβιάσεων και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που γίνεται από ξένα οχήματα οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος. χρειάζεται λοιπόν άμεσα μέτρα να ληφθούν όπως η παρούσα οδηγία για να περιοριστεί η ατιμορρησία των ασυνείδητων οδηγών που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία για να μην συνεχίσουμε να θρηνούμε μια εκατόμβη θυμάτων λόγω των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ε, να πω ότι συμφωνώ με τη ρύθμιση αυτή. Αυτό που θέλω να πω πολύ συγκεκριμένα και που δεν το είπε κανείς μέχρι τώρα είναι ε, το θέμα των σχέσεων με τις υποψήφιες και ενδεχόμενες υποψήφιες χώρες και τις σχέσεις με την Ελβετία. Ε, είναι καλό να ισχύουν όλα αυτά ε, στους 28. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνουν ήδη από τώρα συνομιλίες με όλες τις χώρες όπως Σερβία, Βοσνία και άλλες χώρες αφού και αυτές παίζουν ρόλο καθοριστικό. Εγώ πολλές φορές ε, ε, πιάστηκα οδηγώντας με 90 ενώ το ήταν 80, χωρίς όμως ποτέ να ειδοποιηθώ για πρόστιμο. Ε, επίσης οι χώρες διέλευσης ε, είναι πολύ σημαντικές γιατί εκεί κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές στις διατάξεις μας. Κύριος Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε με μία σύγχυση σε σχέση με τη νομική βάση, η οποία ε, φαίνεται να είναι απαραίτητη. Τώρα εδώ προβαίνουμε στην επικαιροποίησή τη ε, με νέα είδη παραβάσεων, αλλά και ε, με νέε εγγύσει για την προστασία των δεδομένων. Βέβαια, δεν μπορεί να κάνει θαύματα και υπάρχουν πιο βαθιές αιτίε ε, για τα δυστυχήματα όπως ε, το σχάρι ότι οι οδηγοί μπορεί να είναι κουρασμένοι, ότι είναι παλιά τα αυτοκίνητα κτλ. Θα θέλαμε ε, εδώ να αναφερθούμε στο ότι κυριαρχεί στην πρωτοβουλία, στο ότι κυριαρχεί στην πρωτοβουλία το χάρη ότι υπάρχει συνεργασία δημοσίου τομέα, δεν έχουμε καλές υποδομές και πολλές φορές οι οδηγοί αναγκαζόνται να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες οδούς. Φυσικά εδώ είναι απαραίτητη αυτή η οδηγία, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα εις βάθος ζητήματα. Ο κύριος Σόλτες. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνταχθώ και εγώ με τους συναδέλφους που υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Κομισιόν να επιτύχουμε περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους. Η οδηγία είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά περισσότερη κινητικότητα μπορούμε να πετύχουμε μόνο εφόσον εξασφαλίσουμε περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η ανταλλαγή πληροφοριών βεβαίως είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρό. και προκειμένου να συμφωνήσω και με όσους είπαν ότι πρέπει τα στοιχεία να την χάνουν προστασία, τα στοιχεία που ανταλλάσσουμε. Και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό για την ασφάλεια, οι κυρώσεις, οι ποινές που επιβάλλονται. Οι ποινές είναι αποτελεσματικές όταν επιτυγχάνουν τον στόχο. Προκειμένου θα πετύχουμε το στόχο μας Μόνο εφόσον οι ποινέ όντω τελικώ επιβάλλονται. Αυτό είναι και το βήμα που χρειάζεται για να εφαρμοστεί πραγματικά η οδηγία αυτή στην πράξη. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική ευθύνη. Εγκρίνει λοιπόν την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ άλλων σχετικά με τι παραβάσει του κώδικα δική κυκλοφορία. Και μάλιστα πριν το 2016 για να μην προκύψει νομικό κενό, κάτι το οποίο θα αποτελέσει πλήγμα για την οδική ασφάλεια. Χάρη σε προηγούμενε προσπάθειες μειώσαμε τις παραβάσεις που οφείλονται σε ξένου οδηγού. Από εδώ και πέρα, χάρη στον νέο μηχανισμό, θα τιμωρούνται και οι οδηγοί που προπαίνουν σε παραβάσει σε άλλε χώρε. Υπάρχει λοιπόν και νομική ασφάλεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι στον σωστό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Να μειώσουμε κατά 50% του θανάτου στου δρόμου, στου Ευρωπαϊκού δρόμου μέχρι το 2020. θυμίζω μάλιστα ότι η κρίση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλήθους των ατυχημάτων λόγω της ε, χειρότερη υποδομής και λόγω της απουσίας επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε την προτεραιότητα που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει, κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με τα λαθεσμικά όργανα, να προβούμε σε ανταλλαγή στοιχείων και να προβάλλουμε κοινέ εκθέσει για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Επίτροπος Μπούλτ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, καλώ ορίζω πραγματικά αυτή τη συζήτηση. Μου δείχνει αυτό ότι είμαστε ενωμένοι σε ό,τι αφορά το φιλόδοξο αυτό σχέδιο για την τροχιά ασφάλεια. Να επιβεβαιώσω προς ε, όλους σας και όλους μας ε, ότι κάθε θύμα σε τροχαίο είναι ένα θύμα που δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει. Να απαντήσω σε κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Καταρχάς, εν συντομία, τα προσωπικά δεδομένα τα μεταχειριζόμαστε με πολύ προσεκτικό τρόπο και τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις ε, άλλες βάσεις δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς. Υπάρχει πλήρη εγγύηση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Να απευθυνθώ όμως την ανησυχία σας με την οποία συμφωνώ. Φυσικά, αυτό αποτελεί ένα πρώτο μόνο βήμα. Η πραγματική δουλειά πρέπει να γίνει στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί τώρα σε θέματα εφαρμογής. Θα προετοιμάσει μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντας την εφαρμογή της οδηγίας και την ε, αντίκτυπο που θα έχει στην τροχιά ασφάλεια. Όλα αυτά μέχρι το 2016. Αυτή η αξιολόγηση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να κοιτάξουμε περαιτέρω τι θα γίνει, όπως είπατε και κάποιοι από εσάς κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για να καταρτιστούν κοινά πρότυπα για την ασφάλεια στους δρόμους, ε, για τις ε, συσκευές καταμέτρησης, για να εναρμονιστούν οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας και για θέματα πληρωμής ή μη των ε, προστήμων. Αυτό ξέρουμε ότι είναι σοβαρό ζήτημα. Αλλά πρώτα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η τρέχουσα προσέγγιση και τι καρπούς θα αποδώσει ίσως να είναι αρκετά αποτελεσματική ως ε, φόβητρο και να αλλάξει ο κόσμος την οδική του συμπεριφορά. Αν όχι, να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα, όπως μόλις σας εξήγησα. 22 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Έξι ακόμα παραμένουν. Θα συνεργαστούμε μαζί τους στενά για να προχωρήσουμε με τα απαραίτητα βήματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν στην τελική ανάλυση, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για την πραγματικά καλή συνεργασία και προσβλέπω και στη μελλοντική μας συνεργασία για τα θέματα τα οποία δείξαμε. Και φυσικά Προσβλέπω και στην υποστήριξή σα και στην θετική και αισιόδοξη έκβαση της ε, ψηφοφορία αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία η κυρία Γιάννα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπούλτς. Πράγματι υπολογίζουμε στην εμπειρογνωμοσύνη σας και στις ικανότητές σας. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους συναδέλφους για τις πληροφορίες τους ε, και τη συνεισφορά τους γενικότερα. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε στην ασφάλεια την οδική ενέργεια και προσπάθεια και εφόσον υπάρξουν προσπάθειες ε, συντονισμένες θα υπάρξουν αποτελέσματα για τη μείωση των θυμάτων και των νεκρών γενικότερα σε πολλές χώρες μέλη. Πρέπει να εξυγχρονιστεί ο στόλος, Δυστυχώς ε, υπάρχουν πολύ περισσότερα οχήματα από όσο υπολογίζαμε παλαιότερα με πολύ περισσότερα θύματα κάθε φορά. Ε, το θέμα δεν είναι να μειώσουμε μόνο ε, τον αριθμό των νεκρών μέχρι το 2020 αλλά και τον αριθμό των θυμάτων γενικότερα. Οι εμπειρογνώμονες της ITCC μας λέγνε ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των νεκρών στους αυτοκινητοδρόμους ε, με πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή σε, σε ημερήσια βάση ένα σχεδόν ε, ένα αριθμό θυμάτων που φτάνει στο σύνολο των επιβατών ενός μεσαίου αεροσκάφους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την αναθεώρηση της συγκεκριμένης οδηγίας. Αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα θα έχουμε κάνει πραγματικά πολύ πρόοδο για τους πολίτες και για τη βελτίωση του οδικού μας δικτύου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια που κάνουμε έχει σαν στόχο να σώσει ζωές. Τελείωσε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Συγχαρητήρια και στην Επίτροπο κυρία Μπολτσου. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω έναν, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής